Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συνεδρίαση της 17ης ε, Ιουνίου 2013. Και θα ήθελα καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Για αύριο το πρωί υπάρχει μια μικρή αλλαγή καθότι η συνάλφος ε, δεν μπορεί να είναι, ο συνάδελφος Γκάιρ, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι αύριο το πρωί. Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή αλλαγή στη σειρά των θεμάτων. Ε, δύο λεπτά να δω ποιο σημείο θα μπει πριν. Ο κύριος Γραμπάντη λοιπόν θα συζητηθεί το απόγευμα και το σημείο 19 όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα μπει στη θέση του 13, δηλαδή θα γίνει αλλαγή του 13 με το 19. Συμφωνείτε. Εντάξει. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει webstream σε αυτήν την συνεδρίαση. Έχουμε διερμηνία. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες σας γιατί θα υπάρξει και ψηφοφορία. Και να σας πω επίσης ότι η κοινή συνεδρίαση ΛΥΜΠΕ και της δικής μας Επιτροπής θα γίνει Αύριο, 3 με 4. Και φυσικά το θέμα είναι η οδηγία ΠΙΦ. Η συνεδρίαση θα γίνει εδώ, οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα περάσω αμέσως στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων 22, 27, 29 Μαΐου. Έχετε παρατηρήσεις όσον αφορά αυτές, αυτά τα πρακτικά. Δεν βλέπω κανέναν να έχει σχόλια. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε αμέσως και στο σημείο 4. Έκθεση Ντελάγκε. Καταρχήν η εισηγήτρια, επιθυμείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της εφαρμογής της, ε, των υγειονομικών νομοθετικών ε, απαιτήσεων στα νέα κράτη-μέλη είναι αρκετά σημαντικό θέμα και στον δημόσιο και στον πολιτικό διάλογο, γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπάρξει και έχει οθετηθεί νέα νομοθεσία και τα κράτη-μέλη τα οποία γίνονται πλέον μέλη θα πρέπει να ε, συμμορφούνται προς τα κριτήρια αυτά και επομένως να εφαρμόσουν το κεκτημένο. Ήταν ε, νέα η νομοθεσία και επομένως είχαν δυσκολίες και τα παλιά κράτη-μέλη να την ε, υλοποιήσουν και επομένως τα νέα μέλη είχαν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και μεγαλύτερες προκλήσεις απέναντί τους όσον αφορά ακριβώς την υλοποίηση αυτής της νομοθεσίας. Γι' αυτό λοιπόν λοιπόν ε, ε, υπήρξε ε, μία εκτίμηση ότι 117 εκατομμύρια ευρώ από την προενταξιακή βοήθεια θα χρησιμοποιούνται για το θέμα αυτό, δηλαδή την υλοποίηση των υγειονομικών απαιτήσεων σε σφαγεία και αυτά υπό το μέτρο 2 του ΣΑΠΑΡ που αφορά προϊόντα γεωργίας και αλίας. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο έκανε μια ειδική ε, έκθεση έτσι ώστε να δει κατά πόσον τα σφαγεία έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ε, να καλύψουν τις υγειονομικές απαιτήσεις. Διαβάζοντας την έκθεση ήλπιζα ότι θα ε, μπορούσα να έχω τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή πόσα σφαγεία υπήρχαν στην αρχή της διαδικασίας, ποιο ποσοστό σφαγείων κάλυψε ε, τα ε, πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή ήρθε στο επίπεδο της, των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση στα σφαγεία μετά από την χρήση των πόρων Σαπάρα. Όμως αυτό δεν το κατάφερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά να κάνει κανείς μια ασφαλή σύγκριση για το πώς ήταν τα πράγματα πριν τη χρηματοδότηση και μετά και δεν ξέρω τούτη τη στιγμή που μιλάμε και πόσα και ποια είναι τα σφαγεία τα οποία ε, συμμορφούνται ως προς τους ε, κανόνες υγιεινής. Ε, δεν είναι βεβαίως σφάλμα του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος που δεν καλύπτει όλα τα στοιχεία αυτά. Λοιπόν, τι είδε και τι μελέτησε το ελεγκτικό συνέδριο. Τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ποιον επιτήρησε τα χρήματα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν ε, οι ε, πόροι και τελικά εν συμπεράσματι το ελληνικό συνέδριο λέει ότι οι διαδικασίες έχουν ε, ήδη αρχίσει να υλοποιούνται και το σύστημα είναι εντάξει από ό,τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο αλλά βεβαίως ε, εξακολουθεί να διαπιστώνει κάποιες αδυναμίες στα κράτη-μέλη που επισκέφθηκε και στα σφαγεία που επισκέφθηκε. Και αυτό αναφέρω και εγώ στην έκθεσή μου, ας πούμε, για θέματα εποπτείας το ελεγκτικό συνέδριο ε, αναφέρει ότι η αναθεώρηση της ε, Κομισιόν ήταν μερική και όσον αφορά τα προγράμματα εθνικού ελέγχου, τα οποία είναι θεμελιώδου σημασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της ε, νομοθεσίας, βρέθηκαν προβλήματα σε πέντε χώρες μέλη. Όσον αφορά τον σημαντικό τομέα του κτηνιατρικού ελέγχου, επίσης σε πέντε χώρες μέλη υπήρξαν ε, ε, προβλήματα. όσον αφορά τώρα το follow-up, δηλαδή τι θα γίνει με την έκθεση αυτή, την οποία μπορείτε ε, να ε, διαβάσετε και να διαβάσετε και τις απαντήσεις που έδωσε η Κομισιόν. Εξεπλάγει, ε, διότι διεπίστωσα ότι όσον αφορά ας πούμε τον κτηνιατρικό έλεγχο, διαπιστώθησαν αδυναμίες και σε άλλες τέσσερις χώρες, ενώ μόνο μία απήντησε στα ερωτηματολόγια. Επομένως, αναρωτιέμαι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων γνωρίζει πώς έχει η κατάσταση ε, στα ε, άλλα τέσσερα κράτη τα οποία ε, δεν είχαν τους απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους, ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν ποιες είναι οι περαιτέρω επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν. Επίσης, πέραν αυτού μπορείτε να δείτε ποια είναι τα συμπεράσματα στην έκθεσή μου, ποια είναι τα ευρήματα στα οποία αναφέρομαι. Πρέπει να κάνω μια τεχνική διόρθωση γιατί λέω ότι ε, ενθαρρύνουμε την Κομισιόν ε, να ε, κάνει περισσότερους ελέγχους ενώ στο κείμενο αναφέρεται και αναφέρομαι στους νέους τρόπους ελέγχου και στη νέα νομοθεσία ε, στην ε, σελίδα 7 θα πρέπει να αναφερθούν ε, οι νέες προτάσεις που έκανε η Κομισιόν φέτος όσον αφορά τους ελέγχους σε αυτό τον κλάδο. Εν συμπεράσματι λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο είναι ικανοποιημένο γιατί το σύστημα γενικώ δουλεύει ε, θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν ποιες ακριβώς είναι οι αδυναμίες και με ποιο τρόπο ε, προσπαθείτε να τις αντιμετωπίσετε, κυρίως το θέμα του κτηνιατρικού ελέγχου. Παρακαλώ πείτε μου ε, τι έχετε κάνει και ποια συνέχεια έχει δοθεί στις αδυναμίες που διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Και βεβαίως προκύπτει ξανά το ερώτημα το οποίο δεν αφορά μόνο αυτή την έκθεση αλλά είναι πολύ γενικότερο και που αφορά την αποκεντρωμένη δομή με την οποία θέλουμε να εργαζόμαστε. Αλλά όταν αναφερόμαστε στην νομιμότητα, στην νομιμοποίηση μάλλον της ευρωπαϊκής, ε, της ενωσιακής νομοθεσίας, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Εγώ ήλεγξα και ξαναήλεγξα. Ε, η Κομισιόν ακόμα δεν ξέρει ποια και πόσα είναι τα σφαγεία τα οποία χρησιμοποίησαν σωστά τα κονδύλια ΣΑΠΑΡ, πώς ήταν η κατάσταση χρήση πριν στα σφαγεία αυτά και πώς ήταν μετά την χρήση των κονδυλίων αυτών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ε, ψηφοφόρους και οι ψηφοφόροι μας σίγουρα θα θέλουν ε, να ξέρουν ως ε, πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους, θα θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και την εισηγήτρια. Αναφέρθηκε ε, και στο ελεγκτικό συνέδριο και στην Κομισιόν. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Κάρντιφ του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με την απάτη και την Όλαφ και σήμερα ασχολούμαστε με τα σφαγεία. Τρομερές εξελίξεις λοιπόν. Εξαιρετική είναι η εξέλιξη αυτή. Mr. Cardiff, please. Ο κύριος Κάρντιφ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θα σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του συνεδρίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ε, για τα σφαγεία των χωρών που προσχώρησαν στην Ένωση το 2014. Χαιρόμαστε γιατί ε, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας και με την κυρία Ντελάνκη, την οποία και ευχαριστούμε για την εξωτερική αναλυτική της έκθεση. σας αναφέρω το υπόβεθρο της έκθεσης και μετά θα περάσω στα συμπεράσματα. Ξεκινώ με το υπόβαθρο, το ιστορικό. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι οι κανονισμοί για την υγιεινή ε, στα σφαγεία. Είχαμε το πακέτο υγιεινή το 2004, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2006. Σε σύγκριση με τα εφιστάμενα μέχρι τότε κράτη-μέλη που εφάρμοζαν την περιγυνή νομοθεσία της Ένωσης, τα κράτη που προσχώρησαν το 2004 είχαν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις από το νέο πακέτο και τους παρασχέθηκε βοήθεια για τον εξυγχρονισμό των σφαγίων, οπότε και να μπορέσουν να συμμορφωθούν πιο εύκολα με τις νέες απαιτήσεις. Στόχο του δικού μας ελέγχου ήταν να δούμε κατά πόσον η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη που έλαβαν αυτή τη χρηματοδότηση έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφώσουν στα πρότυπα υγιεινής ε, τα σφαγεία τους. Μπορεί αυτό ε, να μην είναι μια τυπική προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν βλέπαμε δηλαδή τόσο πολύ την αποτελεσματικότητα χρήση των κονδύλων, αλλά την υγιεινή, τον κατά πόσον εφαρμόστηκαν οι κανόνες. Κάναμε επισκέψεις σε σφαγεία Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία. Τώρα να έρθω στα βασικά συμπεράσματα. Καταρχάς, θέματα εποπτείας από πλευράς Κομισιών και Κρατών Μελών. Εδώ σχεδιασμό συστημάτων για την εποπτεία των απαιτήσεων ε, υγιεινής από τις αρμόδιες αρχές και τις ήταν μεν, αλλά μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω έλεγχος. Δεύτερο σημείο, η υλοποίηση των απαιτήσεων περί δεν, έχει, δεν είχε εξεταστεί, αναθεωρηθεί πλήρως από την ε, Κομισιόν ε, την στιγμή του ελέγχου Επίσης, βασιστήκαμε στην ε, καταλληλότητα των ελέγχων. Ένα τέταρτο είναι ότι υπήρχαν προβλήματα με το συντονισμό και την τεκμηρίωση ε, και τα προγράμματα και τα αποτελέσματα των ελέγχων των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των απαιτήσεων υγιεινής ασφάλειας τροφίμων, από τους διοικητές, από τους φόρους εκμετάλλευσης. Ναι, μεν υπήρχαν οι κατάλληλε διαδικασίε και πάλι όμω χρειάζεται βελτίωση. Σε πολλά από τα σφαγεία που επισκεφθήκαμε υπήρχαν κάποια ζητήματα υγιεινή, όπω δεν ήταν ε, οι εγκαταστάσει καθαρισμού ε, οι κατάλληλε ή δεν υπήρχε κατάλληλο διαχωρισμό καθαρών από μη καθαρέ ε, περιοχέ. Είδαμε και κάποια προβλήματα με το σύστημα HACCP για την ανάλυση κινδύνων και τα σημεία ελέγχουν. Όπω παραδείγματο χάρη προβλήματα για την καταγραφή ε, ανομαλίων στις θερμοκρασίες. Το σε ό,τι αφορά τα μικροβιολογικά, μικροβιολογική, τη μικροβιολογική δειγματοληψία, οι προθεσμίες δεν τηρούνταν, αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα που διαπιστώσαμε και τέλος και στα συστήματα ανιχνευσιμότητας ε, της προέλευσης του τροφίμου ήταν ένα ζήτημα, ή θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα, δηλαδή η χνηλασιμότητα και με την ε, ταυτοποίηση σφάγιων ε, και ζωοκεφαλαίου υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε δηλαδή πλήρως να βρούμε και ε, την όλη χνηλασιμότητα από το ζωντανό ζώο μέχρι το σφάγιο. Σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση και την εκπαίδευση δεν υπήρχαν ε, κανό, ε, οδηγοί, δεν είχαν εφαρμοστεί, παρότι δεν απαιτείται αυτό βέβαια επισήμω. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα της Κομισιόν Better Training for Safer Food, BTSF. Αυτό έδωσε χρήσιμα, χρήσιμα στοιχεία. Αλλά μπορεί να βελτιωθεί η οργάνωση ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κονδυλίων, να σας πω κάποια πράγματα. Πρώτον, ναι, μεν δεν υπήρξε αξιολόγηση από την Κομισιόν σαφής, αλλά φαίνεται ότι βοήθησαν τα κονδύλια την αναδιάρθρωση των σφαγείων για τη συμμόρφωσή τους προς τα πρότυπα υγείας, αλλά και τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεύτερο, σε κάθε κράτος μέλος που επισκεφθήκαμε, είτε δεν είχε επιτευχθεί η πενταετή σε περίοδο ήταν το κατώτατο όριο, ή τα επίπεδα δραστηριότητα δεν είχαν επιτευχθεί. Και γι' αυτό μειώθηκε η αποτελεσματικότητα τη χρηματοδότηση. Τρει δέσμε συστάσεων έχουμε υποβάλει στην Κομισιόν για να βελτιωθεί η εποπτεία τη της των απαιτήσεων, της τη εκπαίδευση και τη χρήση των κονδυλίων. Όλα αυτά θα τα βρείτε αναλυτικά στην έκθεση. Για να ολοκληρώσω, σημειώνω ότι πρότεινα, πρότεινε η Κομισιόν ε, πρόσφατα μια μείζωνα μεταρρυθμίση απλούστευση τη νομοθεσία περί ασφάλεια τροφίμων και ίσω αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για την Κομισιόν να λάβει υπόψη και τι συστάσει τη έκθεση του συνεδρίου και να τι λάβει σοβαρά υπόψη για να προβεί στι απαραίτητε προσαρμογέ και στις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με τα χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρτιφ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κύριος Μούλτερ. Πολύ σύντομη ερώτηση έχω να κάνω που αφορά την λειτουργία των σφαγείων εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι, τι συμβαίνει, τι κάνει η Επιτροπή, μειώνει ή σταματάει τις ε, επιδοτήσεις και αυτό τι σχέση μπορεί να έχει με την ε, σωστή λειτουργία της αγοράς. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω κανέναν. Η Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο ο κύριος Βαν Έικ από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και ο κύριος Ίος. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Κούνενμπερκ και θα πάρω εγώ το λόγο για το θέμα αυτό. Από μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να σας πω ότι μπορούμε να δεχτούμε όλες αυτές τις συστάσεις. Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες δραστηριότητες και δράσεις. Όσον αφορά τα συμπεράσματα, ο σχεδιασμός αυτού του συστήματος για την παρακολούθηση και την επιτήρηση του συστήματος στα νέα κράτη-μέλη είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί. Συμφωνούμε απολύτως με τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου που λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να ξαναδούμε τον όλο σχεδιασμό του συστήματος για να δούμε αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θέλουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα που διοχετεύονται στην αγορά είναι ασφαλή προϊόντα, ασφαλή τρόφιμα. Οι επίσημοι λοιπόν έλεγχοι θα πρέπει να ενδυναμωθούν και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο έλεγχος αυτός είναι πραγματικά αποτελεσματικός για όλα τα προϊόντα που θα διατεθούν στην αγορά. Κτηνιατρική έλεγχη και άλλοι οι οποίοι θα αυξηθούν και θα ήθελα εδώ να επιμείνω σε τρία σημεία. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κρατημέλη όσον αφορά τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που υπάρχουν, εκδίδοντας ετήσια προγράμματα ελέγχων αλλά και κατευθυντήριες γραμμές. Έλεγχοι οι οποίοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αυξημένη συχνότητα από τις αρμόδιες κτηνιατρικές επιτροπές και υπηρεσίες. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη και θα γίνουν και επιπλέον συστάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύστημα των κρατών μέλων καθότι και να διασφαλιστεί ότι δίδεται συνέχεια μετά από τους ελέγχους, ιδιαίτερα όταν έχουν εντοπιστεί ελλείψεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει λοιπόν να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις της και όσον αφορά το πρόγραμμα για την περισσότερη ασφάλεια στα τρόφιμα, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα ετήσια προγράμματά τους και θα ενημερώνεται τακτικά όσον αφορά την υλοποίηση αυτών. Είναι πολύ σημαντικό οι διάφορες υπηρεσίες να επικοινωνούν, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και ξέρετε ότι υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία εκτελεστική για την υλοποίηση του προγράμματος για μεγαλύτερη ασφάλεια στα τρόφιμα έτσι ώστε πραγματικά να γίνεται ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών σε τακτική βάση. Η βελτίωση του προγράμματος έχει σαν σκοπό καλύτερα αποτελέσματα και αυτό βεβαίως θα μπορέσει να μετρηθεί μέσω αξιολογήσεων και ερευνών που θα γίνουν σε όλα τα κρατημέλη έτσι ώστε να ληφθεί περαιτέρω δράση για να καλυφθούν τυχόν αδυναμίες υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των δράσεων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις του προγράμματος, να υπάρξει μέτρηση των αποτελεσμάτων και υλοποίηση των στόχων. Υπάρχει επίσης και μία σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τους ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα δίκτυο αξιολόγησης για να υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων, εμπειρογνωμοσύνης και πραγματική αξιολόγηση για το 2013. Το πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης έχει απλοποιηθεί και έχει βελτιωθεί. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια Α, συγγνώμη, προηγουμένως ο κύριος Μούλτερ που είχε κάνει μια ερώτηση. Έκανα μια ερώτηση στην Κομισιόν, αλλά εάν δεν σφάλω δεν μου έδωσε απάντηση. Ο κύριος Βαντάικ μήπως θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Ναι, ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Νομίζω ότι οι κανόνες είναι σαφείς. Εάν τα ευρήματα ε, έχουν κάποια επίπτωση στην ε, διατροφική ασφάλεια, τότε ναι, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Ε, εμείς ε, είδαμε τα ευρήματα και δεν έχουν όλα άμεση επίπτωση στην διατροφική ασφάλεια. Μπορεί να παρουσιάζουν ελλειπή συμμόρφωση, αλλά δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην διατροφική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Γιάννης Ευτυχής με την απάντηση. Ε, εάν ε, βεβαίως ε, επιβεβαιωθεί και από την πραγματικότητα θα είμαι ακόμα πιο ευτυχής. Ωραία. Συμπερασματικά σχόλια θέλει να κάνει ο κύριος Κάρντιφ από το ελεγκτικό συνέδριο για να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα κύριε Πρόεδρε. Εμείς δεν είμαστε επιθεωρητές της ασφάλειας τροφίμων και επομένως δεν κοιτάμε το τελικό προϊόν αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν, ε, έχουν βελτιωθεί πολύ περισσότερο ακριβώς και χάρη στη χρήση των ε, ενωσιακών κονδυλίων. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, τα σφάγια ε, την χάνουν σωστότερης επεξεργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα σε επίπεδο υγιεινής είναι πολύ καλύτερο. Ε, βεβαίως εμείς αντιμετωπίζουμε και τα θέματα υγιεινής, αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλά επίπεδα ε, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επομένως δεν είναι σωστό να πούμε εμείς ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα με το τελικό προϊόν αυτό που ξέρουμε από ζητήματα προηγούμενα που σχετίζονται με την διατροφική ασφάλεια, αυτά προκύπτουν όχι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα και μόνο σημείο της διατροφικής αλυσίδας, αλλά ότι ενδεχομένως προκύπτουν από μία σειρά προβλημάτων ε, και ότι κάθε φορά συστηματικά αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας διαπιστώσαμε προβλήματα, εμείς τα αναφέραμε, τα υποβάλαμε στην Κομισιόν έτσι ώστε εκείνη ε, να αναλάβει ε, δράση. Ε, εμείς κάναμε 25 ελέγχους, η κτηνιατρική υπηρεσία κάνει το δεκαπλάσιο κάθε χρόνο και επομένως νομίζω ότι η έλεγχη είναι ικανοποιητική. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, η συνάδελφος Έστεντε Λάγκε. Το συμπέρασμα είναι ότι το θέμα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να συνεχίσει ε, το ενδιαφέρον μας. Έχουμε νέα νομοθεσία και επομένως φαντάζομαι ότι θα ξαναρχίσει η ε, συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι γυρνάμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε ο Γιάνν Μούλτερ για την ασφάλεια των νοοτροφίμων. Βλέπω τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την υγιεινή, ε, κάποια από τα συμπεράσματα αυτά ε, είμαι βεβαία βάσει των παραδειγμάτων που δίνονται ότι οπωσδήποτε υπάρχει επίπτωση στο τελικό προϊόν. Ας πούμε, γίνεται λόγος ε, στην ε, μεταφορά των ε, σφαγίων από βρώμικες προς καθαρές περιοχές. Μάλλον μεταφορά σε καθαρές περιοχές, περνώντας όμως μέσα από βρώμικες περιοχές. Εδώ υπάρχει παραβίαση ενδεχόμενα της νομοθεσίας όσον αφορά την υγιεινή στα σφαγεία. Βεβαίως Ίσως ε, το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα, αλλά τα παραδείγματα τα οποία έχει παραθέσει το ελεγκτικό συνέδριο και το οποίο ε, έχουν προκύψει από τους ελέγχους του οδηγούν σε τέτοιες ε, ε, σε τέτοια ερωτήματα και σε σχέση με την ερώτηση του Γιάν ε, Μιλντερ. τέτοιου είδους προβλήματα ε, που προκύπτουν για προϊόντα τα οποία έχουν βγει στην αγορά περνώντας από τέτοια σφαγεία από σφαγεία δηλαδή που παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα πόσο προβληματικό μπορεί να είναι το τελικό προϊόν η Κομισιόν μπορεί να μας ε, επιβεβαιώσει ότι όσον αφορά τουλάχιστον τον κτηνιατρικό έλεγχο αυτά τα, ε, ε, σε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία επισκέφθηκε και στα οποία υπήρξαν ελλείψεις για αυτές τις τέσσερις από τις πέντε χώρες μέλη έγιναν κάποια βήματα, ε, η, παρακολουθεί η Κομισιόν την κατάσταση, τα κράτη-μέλη έλαβαν μέτρα τα οποία έχουν οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό να μας πει η Κομισιόν. Και επίσης ε, η τελική παρατήρηση ε, ήταν ακριβώς ότι ε, ξεκινάμε τώρα την σύνταξη νέας νομοθεσίας και επομένως ε, πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας. Ε, και επομένως ερώτηση, τι μπορεί να μας πει το ελεγκτικό συνέδριο, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι επίσημοι έλεγχοι. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα έτσι ώστε να είναι πιο σωστές οι νέες προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος και θέλει να πάρει το λόγο. Ja mam dalej brak Έχω την εντύπωση <clears throat> ότι δεν είχα αρκετέ πληροφορίε όσον αφορά τι διαδικασίε. Τι ακριβώ έλεγξε το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά τα σφαγεία. Σε ποια βάση, αν θέλετε, μπορεί κανείς να τεκμηριώσει αυτές τις συστάσεις που προτείνετε; Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Και αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο, ότι κάνετε κάποιες γενικεύσεις των στοιχείων που έχετε. Ήταν τόσο γενικά αυτά που μας είπατε, που πραγματικά θα μπορούσε κανείς να τα συμπεριλάβει σε κάθε περίπτωση ε, έκθεσης. Ό,τι και να ήταν, αν θέλετε, ο έλεγχος. Ξέρω βεβαίως ότι υπάρχει θέμα κόστους, ότι η μεταρρύθμιση μιας νομοθεσίας, ρυθμίσεων είναι εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία. Εγώ είμαι μέλος και της ε, Επιτροπής Γεωργίας και ξέρω πώς περνάει κανείς από τις προτάσεις στην πρακτική. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ γενικά αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή. Όπως είπε και η συγκήτρια, είμαστε Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά δαπανήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά εάν υπάρχει υλοποίηση των στόχων, εάν υλοποιείται ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Αυτή η προσέγγιση μας ενδιαφέρει. Η κυρία Ντελάγκε λοιπόν μίλησε για δύο πράγματα. Ο έλεγχος, η ποιότητα των τροφίμων που βγαίνουν από τα σφαγεία και εάν τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο έχουν διατεθεί. Και βεβαίως τι μπορεί να γίνει αν η απάντηση είναι αρνητική. Okay, I think I will respond on behalf of... Να απαντήσω, βέβαια από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και επικεντρώθηκα στα στήματα της υγιεινής. Έγινε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τους ελέγχους. Θα δώσω το λόγο μετά τους αρμόδιους για τη Γεωργία συναδέλφους μου που θα σας μιλήσουν για το σκέλος της χρηματοδότησης. Να επιβεβαιώσω λοιπόν ότι μετά τον λογιστικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου στα πέντε κράτη-μέλη το ένα απάντησε, τέσσερα όχι. Αυτά τα κράτη βέβαια εξολογήθηκαν από την υπηρεσία τροφίμων, την κτηνιατρική και κτηνιατρική FVO. Και μετά έγιναν και κάποιες συστάσεις και υπάρχει μια παρακολούθηση, μια συνέχεια στις δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη αυτά για να εφαρμόσουν πλήρως την νομοθεσία περιγυρνής. Αυτές τις εκθέσεις ε, μπορείτε να τις βρείτε, είναι διαθέσιμες. Δεν εντοπίστηκαν σε αυτές ε, μείζωνα ζητήματα υγιεινής ασφάλειας τροφίμων, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όπως γίνεται συνήθως με τους ε, ελέγχους του ΕΦΙΟΥ, e Φυσικά αφορούν και το σκέλος της υγιεινής, έγιναν οι αξιολογήσεις και υπάρχουν και σχετικές εκθέσεις. Για το δεύτερο ερώτημα θα προτιμούσα να δώσω το λόγο σε συνάδελφους με τη ΓΑΜΑ Άγκρη, οι οποίοι θα μπορούσαν να απαντήσουν πιο συγκεκριμένα για τα ζητήματα της ε, χρηματοδότησης που δόθηκε για την ε, συμμόρφωση προς τις απαιτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή ή η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχει ορίσει μία περίοδο πενταετούς παρακολούθησης αφού δόθηκαν τα κονδύλια για αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως κάποιες χώρες ζητούν επτήσιο έλεγχο έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά τηρούνται οι προδιαγραφές για τα σφαγεία τες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν λοιπόν έλεγχοι όσον αφορά τη συμμόρφωση αυτών των εγκαταστάσεων από τους ελεγκτές μας. Okay. Äh, Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο μετά από αυτές τις απαντήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα περάσουμε στο επόμενο. Πρόκειται για την ειδική έκθεση. Στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βεβαίως από το ελεκτικό συνέδριο έχουμε εδώ μαζί μας τον Άσα Ούπεργκίτε. Θα σας δώσω το λόγο. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και σας δίνω το λόγο. Ah, Moment. Yes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Έγινε ο έλεγχος 121 για τον συγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σκοπό σκοπός μας ήταν να δούμε εάν ο εξυγχρονισμός αυτός ε, έχει επιτευχθεί και ώστε να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι που βεβαίως ζητήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη και το πιο βασικό θέμα ήταν τα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί, 11,1 δις, 11% δηλαδή των δαπανών για τις ε, ε, γεωργικές δαπάνες για τις επάνες για την Ήπεθρο και βεβαίως ε, εδώ έχουμε μια ολόκληρη σειρά σχεδίων για την Ήπεθρο που αφορούν αυτά τα προγράμματα. Τα ειδικέ ανάγκες των κρατών μελών, καθώς και οι προτεραιότητες όπως η καινοτομία, η διαφοροποίηση είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Έχουμε θέσει ειδικού στόχου με σκοπό βεβαίω να αντικατοπτριστούν οι προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ειδικέ ανάγκε των κρατών μελών με στόχους επιλεξιμότητας και κριτήρια για να επιλεγούν τα καλύτερα προγράμματα, βιώσιμα προγράμματα και έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι υπερβολικοί κίνδυνοι που εμπεριέχονται. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας εδώ και τις ε, διάφορες δαπάνες που είναι προαπαιτούμενα για αυτόν τον εξυγχρονισμό. Και εδώ έχουμε τον πολύ συγκεκριμένο στόχο να υπάρχει καλή χρήση αυτών των κονδυλίων. Οι στόχοι αυτοί βεβαίως είναι κάτι που έγινε μετά από μια συγκεκριμένη θέση προτεραιοτήτων. Μόνο δύο κρατημέλη είχαν πολύ συγκεκριμένους ε, στόχους και προτεραιότητες, τρεις είχαν συστήματα προτεραιοτήτων πολύ περιορισμένα. Πρόκειται για περιορισμένα και αδύναμα συστήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα η χρήση των κονδυλίων να μην γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, λέγξει και εγκρίνει προγράμματα για την ε, ανάπτυξη της υπέτρου βάση συγκεκριμένων κριτήριων. Το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στην Επιτροπή να καθορίσει κατά πόσο αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν. Επίσης υπήρχε ελλειπής ε, θέση προστεραιοτήτων και στόχων, κάτι που οδήγησε σε περιορισμένη επιπλέον χρηματοδότηση όσον αφορά τους υγειονομικούς ελέγχους. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό το έχει εντοπίσει το ελεγκτικό συνέδριο, να δούμε που υπήρχαν προγράμματα με βιωσιμότητα, οικονομική βιωσιμότητα, και το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι το κοινό πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό όσον αφορά τα αποτελέσματα και όσον αφορά την βιωσιμότητα των στόχων, των επενδύσεων, καθώς και την αξιολόγηση η οποία δεν έγινε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού 121. Καταρχήν, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθετικό έργο, το οποίο να λαμβάνει υπόψη του με σαφήνεια τις απαιτήσει και τις ανάγκες των κρατών μελών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτές οι απαιτήσει υλοποιούνται και ότι από τη στιγμή που τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου αποφασίζονται, λαμβάνονται υπόψη οι ε, διάφοροι στόχοι και τα κριτήρια. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθούν οι προτεραιότητες στο εσωτερικό αυτών των υγειονομικών ελέγχων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νομοθεσία για να συμμορφωθούν αυτές οι διαδικασίες προς τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικά αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση και αυτή να διευκολυνθεί. Τέταρτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν ε, αποτελεσματικές διαδικασίες οι οποίες ε, να λαμβάνουν υπόψη τους με αναλογικό τρόπο τους κινδύνους. Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις δαπάνες των επενδύσεων έτσι ώστε να μπορούν να μπουν στους στόχους της επιλεξιμότητας. Οι προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου λαμβάνουν υπόψη της όλα αυτά τα δεδομένα και προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις συστάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τέλος, το ελεγκτικό συνέδριο προτείνει να συσταθούν κριτήρια κόστος οφέλους έτσι ώστε να μπορέσει να μετρήσει στην επόμενη αξιολόγησή της και την καινοτομία. Ο ρόλος της διαχείρισης είναι να προτείνει αυτά τα κριτήρια. Παρόλα αυτά, το ελεγκτικό συνέδριο θα ελέγξει στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης και ελέγχων αυτήν την ύπαρξη τέτοιων ε, κριτηρίων καθώς και την ύπαρξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολισμού για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική παρουσίαση την κυρία Μπουτμπεργκητέ και πράγματι είναι πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Το πλαίσιο ήταν πολύ θετικό. Είναι μια σημαντική έκθεση αυτή, δεν λαμβάνοντας υπόψη το πόσο λεπτό θέμα είναι τα μέτρα, ε, αγροτική ανάπτυξη και ΚΑΠ, και γεωργική πολιτική. Εδώ μιλάμε για την πρώτη βέβαια, είναι το πρώτο θέμα, η ανάπτυξη της υπέτα, αγροτική ανάπτυξη και υπάρχουν διάφοροι πυλώνες. Σημαντικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων, την διαχείριση του εδάφους, ε, τη διατήρηση των τοπίων κτλ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, πρόσωπος ε, του Εκτικού Συνήθου μας παρουσίασε το μέτρο 121 που σχετίζεται με τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εδώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι εύστοχα τα συμπεράσματα και Ακριβώς επειδή αυτή η ανάπτυξη πέτρου είναι ένας νέος πυλώνας και έχουμε τις ε, διατάξεις που εφαρμόζονται πλέον για τον έλεγχο και τα λοιπά και έχουμε και το κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές. Θα έχουμε λοιπόν έναν ε, σταθερό συμπαγή μηχανισμό που δίνει αξιοπιστία και καλά αποτελέσματα ελέγχου και αξιοπιστία. Στην περίπτωση της αγροτικής ανάπτυξης δεν υπήρχε, έπρεπε να, καταρχάς να δημιουργηθεί και κατά δεύτερον αυτός ο μηχανισμός να ενισχυθεί. Και αυτό γιατί είναι ανάγκη μεταξύ άλλων να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα και τον μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης, αυτό το κοινό πλαίσιο ελέγχου και παρακολούθηση για τα μέτρα περί ανάπτυξη πέτρου. Μιλάμε λοιπόν για το μέτρο 121, 11,1 δις περίπου είναι το ποσό, δεν είναι βέβαια και το πιο τεράστιο ε, ποσό, αλλά είναι σημαντικό. για την επίτευξη των ε, στόχων. Συμφωνώ με όσα είπε η πρόσωπος του Ελληνικού και τα συμπεράσματα, πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα και το πλαίσιο ελέγχου και επακολούθηση αλλά κατά πόσο πρέπει να πετήσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μια ομοιογενοποίηση των δεδομένων που τροφοδοτούν το σύστημα και σε ό,τι αφορά τους δείκτες αυτοί οι δείκτες κατά την άποψή μου θα πρέπει να βοηθούν στο να γίνει μια συγκριτική ανάλυση και να καταλήξουμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα ελέγχου και αξιολόγηση. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε τη διασπορά, αν μπορώ να το πω έτσι, και σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις και σε ό,τι αφορά το σκέλος της εφαρμογής. Υπάρχει εδαφική πυκλομορφία, άρα αυτό απαιτεί ευελιξία. Αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει να έχουμε καταγερματισμό και διασπορά. Γιατί έτσι θα περιοριστεί η δυνατότητα δράσης. Συμφωνώ επίσης ως προς το ότι πράγματι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανομοιογένεια και ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προτεραιοτήτων. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει η αξιολόγηση με κάποιο ομοιογενή τρόπο. Είδαμε και το χρονοδιάγραμμα και σε κάποιες χώρες, στη Ρουμανία για παράδειγμα, δεν μπόρεσαν να δώσουν όλα τα στοιχεία όταν τα του ζητήθηκαν. Ε, άρα έδειξαν αρνητικές επιδόσεις, ενώ τελικά ε, φάνηκε στο τέλος ότι είχαν ένα καλό σύστημα, απαιτητικό σύστημα, και δείκτες, οπότε το αποτέλεσμα το τελικό ήταν πολύ πιο θετικό από άλλα εδάφη που αξιολόγησε το ελεκτικό σεντρίο, Όπως Βάδη Βιτεμβέργη, Καταλωνία, όπου είπαμε ότι εκεί πρέπει να είναι αρκετά συμβατά μεταξύ τους τα κριτήρια και οι δείκτες, αλλά ε, δεν υπήρχε αυτό. Αποτέλεσμα είχαμε και απρόβλεπτες συνέπειες αλλά και τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τον εξυγχρονισμό των λειτουργικών συστημάτων των εκμεταλλεύσεων αυτών. Έχει αποδειχθεί ότι ανεξάρτητα από την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων και υποβολητημάτων και αξιολόγησης θα πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δηλαδή έχουν εξεχρονιστεί και σε μεταλλεύσεις, αλλά κάτι άλλο που βοηθά είναι και η διαγενειακή ε, αλλαγή. Το πέρασμα δηλαδή από ε, τη μια γενιά στην άλλη της σκητάλης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. la redundancia sobre cómo está aplicando. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένε παρατηρήσει ω προ τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία του ελληνικού συνεδρίου, αλλά θα επιμείνω σε κάτι. Κάποιε φορέ έχουμε κάποιε αντιφάσει. Δηλαδή, το ελεγκτικό συνέδριο μα εξηγεί και λέει ότι είναι λογικό να υπάρξει εξυγχρονισμό όταν έχουμε αγορά μηχανημάτων, όταν έχουμε επενδύσει. φυσικά λένε είναι λογικό ότι υπάρχει εξυγχρονισμό. Και μετά όμως μας λένε ότι ναι μεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει εξυγχρονισμό. δεν εκπλήττω στα τα κριτήρια για καινοτομία. Ζητώ λοιπόν να, να μου πείτε το εξή, να μου διευκρινίσετε για να έχουμε και διαφάνεια. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησε το ελεγκτικό. Διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιε αντιφάσει στην έκθεση. Γιατί εκεί που είδαμε ε, ότι σαφώς ε, τα συστήματα δεν ήταν αποτελεσματικά όπως περίπτωση του Λουξεμβούργου ή της Πολωνίας η περίπτωση επίσης ήταν μια από αυτές βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις Γι' αυτό, για να είμαστε σαφείς περισσότερο και για να μπορέσει να εφαρμοστεί και πιο σωστά στο μέλλον αυτός ο μηχανισμός, θέλω να μου πείτε ακριβώς πού πιστεύετε ότι πρέπει να θεσπιστούν αυτά τα κριτήρια και ιδίως περί κόστος ωφέλους. Γιατί Λέμε από την αρχή, ναι, να υπάρχουν επενδύσεις, νέα συστήματα διαχείρισης, νέα μηχανήματα, νέος εξοπλισμός. Αυτό σίγουρα συνεπάγεται συγχρονισμό, αλλά δεν συνεπάγεται καινοτομία. Δεν ξέρω. Ποια είναι τα κριτήρια για την καινοτομία τα οποία εφαρμόζει το ελεκτικό συνέδριο και κάτι άλλο που θέλω να αναρωτήσω. Ε, χρησιμοποιήσατε διαφορετικά εδαφικά στήματα. Δηλαδή για την Ισπανία, Καταλωνία, για τη Γερμανία, Βάδη, Βερτεμβέργη, εδάφη, περιοχές που δεν είναι και αντιπροσωπευτικά πόλη. Εντάξει, για το Λουξεμβούργο είναι πιο μικρό, αλλά πια σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Για τη Ρουμανία εκεί εμφανίζεται ολόκληρη χώρα, όχι μια περιοχή της χώρας. Μήπω μπορείτε λοιπόν να μα δώσετε πιο πολλά στοιχεία για τα κριτήρια, γιατί κάνοντα τη συγκριτική ανάλυση πώ επιλέγουμε την Καταλωνία για να ε, εκπροσωπήσει όλη την Ισπανία, για παράδειγμα, για τον εξεχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα είναι αλλιώς ε, το φωτογραφικό στιγμιότυπο αν χρησιμοποιήσουμε την Καταλωνία σε σχέση με το αν χρησιμοποιούσαμε την Εστρεμαδούρα ή κάποια άλλη περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από το τελικό Συνέδριο να μας κάνει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση και με το μέλλον, για να μπορέσουμε δηλαδή και στο μέλλον να μετρήσουμε καλύτερα. Πώς να το πω. Το ενδιαφέρον μας, το συμφέρον που έχουμε και εμείς να έχουμε σαφείς απαντήσεις από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και θα περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, η κυρία Ντελάνγκη. Να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε η συγγήτρια, τι γίνεται δηλαδή με τα ε, κριτήρια επιλογής και πώς ε, ε, πώς έκανε την επιλογή η Κομισιόν, ε, γιατί ξέρουμε ότι δύο ομάδες ε, έπιαναν τα κριτήρια, δύο καθόλου και υπήρχε και μία ενδιάμεση ε, ομάδα. Επίσης, στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης υπαίθρου έχει προταθεί από την Κομισιόν να υπάρξουν και επιπλέον στόχοι ας πούμε, ε, στην διαχείριση των υδάτων, την κλιματική αλλαγή και την βιοπικιλότητα. Πόσο μακριά πάει η Κομισιόν και κατά πόσον καλύπτονται και κάποια από τα άλλα κριτήρια σε αυτούς τους νέους τομείς. Γιατί μπορεί, ας πούμε, κάποια μέτρα να είναι καλά για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων αλλά να είναι πολύ επιβλαβή για την κλιματική αλλαγή ας πούμε. Ε, στα πλαίσια της ε, κοινή γεωικής πολιτικής ελέγχει η Κομισιόν όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματικά win-win κατάσταση όλα αυτά τα επιπλέον κριτήρια δηλαδή καλύπτονται όσον αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και άλλες. Μπορεί να μας δώσει η Κομισιόν κάποια παραδείγματα σχετικά με το πώς από τα ε, ε, κονδύλια που έχουν χρησιμοποιηθεί πηγαίνουν ακριβώς σε αυτήν την διτή πρόοδο, την win-win κατάσταση και πόσα είναι τα κονδύλια τα οποία αφορούν παραδοσιακές μορφές ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ο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 αλλά και επί του κόστους. Το γεγονός ότι κάποιος αποφασίζει να εξυγχρονίσει μια γεωργική εκμετάλλευση, τουλάχιστον να κοιτάξει να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τουλάχιστον αυτό. Επίσης, τα κονδύλια για τον εξυγχρονισμό θα πρέπει να ειστρέουν κατευθείαν για τους δικαιούχους, να φτάνουν στους δικαιούχους. Έχω λοιπόν ένα σχόλιο να κάνω. Όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης, ε, αγροτικής ανάπτυξης και όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού, θα ήθελα να δούμε κατά πόσο είναι στοχευμένη η κατανομή των κονδυλίων και ποιες οδηγίες ισχύουν εδώ. Οι οδηγίες για την γεωργία, αυτές που περνάνε δηλαδή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Δεν προσπαθώ να προσάψω σε κανέναν κάτι που δεν έγινε σωστά. Προσπαθώ να καταλάβω. Η συγγήτρια ανέφερε τα θέματα αυτά και θα ήθελα να μου πείτε η αύξηση της ανταγωνιστικότητας έχει σχέση με την επιφάνεια που διαθέτει ένας αγρότης. Γιατί εδώ πολλές φορές βλέπουμε ότι αλλιώς εξυγχρονίζεται μια μεγάλη επιφάνεια, μια μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση και τελείως διαφορετικές είναι οι ανάγκες των μικρών γεωργών. Είναι πολύ δύσκολο, παραδείγματο χάρη, κάποιος να αγοράσει κάποια πολύ σύγχρονα μηχανήματα από τη στιγμή που δεν ανταποκρίνονται στην καλλιέργεια και στην επιφάνεια που διαθέτει. Ίσως θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να μπορεί να στοχεύσει πιο συγκεκριμένα τον εξυγχρονισμό που είναι απαραίτητος για την ε, γεωργική του εκμετάλλευση. Δηλαδή υπάρχει ο βασικός εξοπλισμός και κάποιες άλλες απαιτήσεις και ανάγκες ε, που δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όλες τις επιφάνειες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτές τις ιδιαιτερότητες αλλά αυτό έχει άμεση σχέση και με το μέγεθος, με την επιφάνεια. Οι μεγάλες, παραδείγματο χάρη γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ε, ε, Ολλανδία έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες από μια γεωργική εκμετάλλευση στην Πολωνία ή στην Ρουμανία. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η βάση, ο βασικός εξοπλισμός που πρέπει να εξυγχρονιστεί και μετά βλέπουμε και όλα αυτά προϋποθέτουν και απαιτούν διαφορετικά κριτήρια και διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε εδώ να έχουμε μια ενιαία ε, και εναρμονισμένη προσέγγιση από μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Ας κοιτάξουμε, επαναλαμβάνω, το βασικό σχέδιο εξυγχρονισμού και όχι τις πολύ εξειδικευμένες ε, μηχανές, τις οποίες είναι, αν θέλετε, πολλές φορές ανίκανοι πολλοί γεωργοί να χρησιμοποιήσουν δεδομένες της ε, επιφάνειας που διαθέτουν και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να έχει ζητήσει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ο Χωσέ Μανουέλ Σούζα και ο κύριος Χανιώτης. Ποιος θα πάρει το λόγο. <clears throat> <clears throat> Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και την εισηγήτριά του για την ε, εργασία τους, τις συστάσεις τους, έτσι όπως τις παρουσίασε η εισηγήτρια. Εμείς ευθυγραμμιζόμαστε με τις ε, προτάσεις όσον αφορά και το μέλλον και όσον αφορά την επίτευξη στόχων και τις σχέσεις κόστους-οφέλους για τα, για τα δημόσια κονδύλια. Συμφωνούμε λοιπόν Αλλά βεβαίως ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήδη, ήδη ε, καταβάλλονται προσπάθειες ε, τώρα, στην παρούσα περίοδο. Η σύσταση 1, αβ, θέλω να πω επ' αυτού ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί, τρόποι στόχευσης της ε, βοήθειας. Υπάρχουν βεβαίως τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά ε, υπάρχουν και άλλα κριτήρια ε, τύπος επένδυσης, τύπος δικαιούχου, εντατικοποίηση, βαθμός εντατικοποίησης κτλ. Το κάθε πρόγραμμα βασίζεται σε κάποια στρατηγική. Στο μέλλον η στρατηγική προσέγγιση θα ε, επιταθεί ε, και επομένως θα υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική η οποία θα σχετίζεται με τους στόχους της ε, περιφέρειας και της χώρας ανάλογα αν μιλάμε για εθνικό προγραμματισμό ή περιφερειακό προγραμματισμό. Επίσης, στην ενισχυμένη στρατηγική προσέγγιση ε, θα ταυτοποιούνται οι ανάγκες και θα προτείνονται οι απαραίτητες επενδύσεις, αυτές δηλαδή που χρειάζονται έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερα ο στόχος που έχει τεθεί. Βεβαίως ε, πολλά εξαρτώνται από τον βαθμό ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής. Δηλαδή κάτι που είναι καινούριο για μία περιοχή μπορεί να είναι παλαιό και γνωστό για κάποια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα πρέπει κάθε φορά να επιβεβαιώνεται η κατάσταση. Επίσης, τα πόσο αναφορά τα κριτήρια επιλογής, ε, ναι, βεβαίως ότι οι νέες προτάσεις ε, θα επιτείνουν την ανάγκη για πιο στοχευμένα κριτήρια επιλογής. Για την ε, ώρα να θυμίσω ότι έχουμε το share management και κατά αυτή την έννοια το κράτος ε, ε, μέλος θα πρέπει να δώσει μία εκ των προτέρων εξάντε αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ε, του προγράμματος που προτείνει για μια περιφέρεια ή για μια χώρα. Στο μέλλον ε, ξέρετε ότι η στόχευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα καθορίζουμε περισσότερο στόχους βάσει έξι προτεραιοτήτων και για κάθε προτεραιότητα τρεις ε, focus areas. έτσι ώστε η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε να είναι καλύτερα στοχευμένη και να αρμόζει καλύτερα στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στην νέα νομοθεσία και μάλιστα στο άρθρο 18 της νέας πρότασης δίνεται η δυνατότητα καλύτερης στόχευσης λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες της εν λόγω περιοχής και δίνεται τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν καλύτερα και από τη δική μας πλευρά να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα την ε, χώρα μέλος. Οι στόχοι προκύπτουν από συγκεκριμένους συντελεστές και παραμέτρους. Eh, και στη σύσταση 2 μάλιστα ε, η αναφορά λέει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ε, η εποπτεία. Ναι βεβαίως συμφωνώ αλλά θα ήθελα να σας πω τούτο. Ήδη υπάρχει ένα πλαίσιο κοινής αξιολόγησης και αυτό είναι από τα πιο αναπτυγμένα Ε, όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία ας πούμε. Βάσει και του κανονισμού 6019 υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μην είναι τέλειο, βεβαίως πρέπει να ε, βελτιωθεί περαιτέρω, αλλά παρόλα αυτά παρόλα αυτά έχουμε μια εμπειρία η οποία μας δίνει την ε, ε, δυνατότητα να κάνουμε τον ενδιάμεσο έλεγχο και την ενδιάμεση έκθεση ε, που βασίζεται σε κάποιες ενδείξεις, έναν αριθμό δικτών δηλαδή που μπορεί να μην μας δίνει τα τέλεια στοιχεία, αλλά τουλάχιστον μας προειδεάζει για την κατάσταση. Η περίοδος αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί της πρώτης ε, ε, αναθεώρησης. Ε, το 15 θα είναι αυτό και βεβαίως τότε θα κάνουμε και την εξπόστα, την εκ έκθεση αξιολόγησης. και όλα τα στοιχεία θα μπορούν να επαληθευθούν πλήρως. Επομένως, κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, αυτό το έχουμε ήδη ε, και ε, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την αξιολόγηση και την εποπτεία. Ε, πολλές προσπάθειες καταβάλλονται για να συνεργαστούμε και με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε όλοι να έχουν καλύτερη επίδοση για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Να πω και δύο λόγια όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα που θεωρεί στη σύσταση 4 το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Βεβαίως και στο μέλλον τα μέτρα και η οικονομική δραστηριότητα θα διασυνδεθούν με business plans, με επιχειρηματικά ε, σχέδια. Για μία ακόμα φορά να πω ότι και εδώ βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Από τη μία πλευρά την ε, απλούστευση. Δεν θέλουμε επιπλέον ε, διοικητικό κόστος ε, για τις χώρες. Και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά τα οποία μας υποχρεώνουν να είμαστε πιο ευρωματικοί όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν την σωστή αξιολόγηση. Προσπαθούμε να εξεύρουμε λοιπόν την σωστή ε, ισορροπία έτσι ώστε να δίνουμε και τη σωστή πληροφόρηση προς τις ε, χώρες μέλη. Και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει, ε, θα, θα, θα περάσουμε αυτή τη διαδρομή έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλό αποτέλεσμα η ενίσχυση των στόχων που ανέφερα ε, και τα business plans τα οποία θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα είναι ένα πολύ σωστό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα ε, βοηθήσει έτσι ώστε να μειωθούν ε, οι ενεχόμενοι κίνδυνοι. Στην παρούσα περίοδο και στη διαδικασία ευθυγράμμισης ε, της ε, νομοθεσίας που έχουμε μπροστά μας. Ε, σε αυτές τις διαδικασίες, λέω, οπωσδήποτε θα πρέπει να βρούμε νέες πειθαρχίες όπου θα υπάρξει δυνατότητα επιλεξιμότητας μετά τον καθορισμό των, των πιστώσεων πληρωμών, συγγνώμη, υποχρεώσεων και επίσης έλεγχος εκ των υστέρων μετά την ε, ε, απόφαση επιλεξιμότητας. Νομίζω ότι με τα δύο αυτά μέτρα κάλυψα, αν όχι όλες, αλλά τουλάχιστον τις περισσότερες παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Και βεβαίως ε, με χαρά θα συνεχίσω τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε στο μέλλον τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής μας να είναι όλο και πιο σωστά και πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Άλλα σημεία τα οποία θέλετε να εγείρετε. Διαφορετικά να ξαναδώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο, εάν βεβαίως επιθυμεί η εκπρόσωπός του να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντες για τα ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα τα οποία έθιξαν. Να ξεκινήσω από τα ερωτήματα της εισηγήτριας. Πρώτον όσον αφορά την στόχευση και τα κριτήρια επιλογής. Η νέα νομοθεσία θα θέσει νέους στόχους για τα μέτρα. Και αυτό βεβαίως είναι πολύ γενικό. Μετά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία ε, θα καθορίσουν πλήρως ε, τους ε, στόχους με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν σαφώς τις ανάγκες τους και τις προτεραιότητες τους. Τα κράτη-μέλη στα πλαίσια ενός σαφούς και, εξειδικευμένου, και εξειδικευμένα στοχευμένου προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου μπορούν ε, να καθορίσουν ε, το πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει συγκεκριμένες κατηγορίες ε, δικαιούχων διαφοροποιημένου ποσοστά ε, βοήθειας ανάλογα με το, τα προγράμματα κλπ. Επίσης συγκεκριμένα κριτήρια ε, για τον καθορισμό αυτών των προγραμμάτων που περισσότερο συμβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων και επίσης ε, τα ε, ε, προγράμματα τα οποία περισσότερο αναφέρονται σε μείωση των κακών επιπτώσεων, μείωση του κενού βάρους κτλ. Εμείς στη δικιά μας έκθεση και μάλιστα στην παράγραφο 26 και στην παράγραφο 27 και στην παράγραφο 28 άλλωστε δίνουμε ε, κάποια παραδείγματα σε σχέση και με το πλαίσιο 2, box 2 έτσι ώστε όλα τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουμε βρει ε, στις ε, χώρες μέλη να αναλυθούν και να επιτευχθεί καλύτερα. Πούμε για την Ουγγαρία. Λέμε ότι οι αρχές έχουν κάνει διαγωνισμούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα άρδευσης κλπ. Και βεβαίως οφείλει να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα από τη στιγμή που το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να κάνει αυτόν τον έλεγχο και τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, εφάρμοσαν τα κριτήρια από τη δική τους πλευρά τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορές κατά την άποψή μου από τα δικά μας κριτήρια ελέγχου και ε, των κριτηρίων επιλογής στα ίδια τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία μπορούν καλύτερα να στοχεύσουν τα τον σκοπό των προγραμμάτων και μπορούν να βοηθήσουν ε, ε, καλύτερα τις περιφέρειες ή τις χώρες ανταποκρινόμενες σωστότερα στις ανάγκες τους. Η κυρία Γιάλα Σέντερ είπε ότι βλέπει κάποιες ε, αμφισημίες στην έκθεσή μας. Εγώ δεν τις βλέπω τις αμφισημίες αυτές. Απλώς κάποιες διαφορές ε, είναι αναπόφευκτες. Ε, βελτιώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση όταν δαπανώνται χρήματα για νέα εργαλεία και νέα μηχανήματα. Ωστόσο, τα ενωσιακά κονδύλια θα είχαν επιτύχει καλύτερα το στόχο τους εάν η στόχευση της χρήσης των χρημάτων αυτών ήταν καλύτερη. Και νομίζω ότι αυτό το αναφέρουμε ρητά στην έκθεσή μας. Όσον αφορά τώρα την ε, επιλογή των κρατών μελών και τη διάρκεια του ελέγχου. Ο έλεγχος αφορούσε 10 χώρες, 7 εκ των οποίων ε, δέχτηκαν επιτόπου επισκέψεις. Η επιλογή των κρατών μελών εξαρτάται πρώτα απ' όλα από το επίπεδο δαπανών ε, των ε, κρατών μελών ή της ε, συγκεκριμένη περιφέρειας σε κάποια χώρα μέλος. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το κράτος μέλος, όπως ας πούμε η Πολωνία, μπορεί να έχει προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης συνολικής, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν κάτι τέτοιο. Το ελεγκτικό συνέδριο προσπάθησε να λάβει υπόψη το ελεκτικο συνεδριο προσπαθησε να λαβει υποψη το τη γεωγραφική διάσταση και εν τέλει μια εξισορροπημένη κάλυψη παλαιών και νέων κρατών μελών έτσι ώστε να υπάρξει ε, σωστή σύγκριση και έτσι ώστε το ελεγκτικό συνέδριο να μπορέσει να εξάγει σωστά συμπεράσματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνει σωστές προτάσεις. Δεν νομίζω ότι έχω τίποτα άλλο να πω. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκούτε. Η συγγήτρια θέλει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και για τα σχόλια. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το οποίο σχολίασα και εγώ Είμαστε και στη νέα φάση προγραμματισμού. Θα πρέπει, μας εξήγησε η Κομισιόν να, ε, να λάβουμε υπόψη μας και την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, να εκμεταλλευτούμε το διάλογο που έχουμε και τις συστάσεις της Επιτροπής για να βελτιώσουμε τα προτινόμενα μέτρα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και το είπαμε. Όχι μόνο για τη διατήρηση και τον εξεχρονισμό των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και γιατί θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα απασχόληση και μάλιστα ποιοτική. για την ευέλτιστη διαχείριση της, ε, των εδαφών. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ε, την ε, διαγενειακή αλλαγή. Βέβαια δεν επιμένω γιατί έτσι θέλω, απλά γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι εκθέσεις του ελληνικού συνεδρίου να επηρεάζουν, να έχουν έναν αντίκτυπο και έχουν αντίκτυπο. Και για να κάνει τις απαραίτητες τροποποίησεις κομισιών, αλλά και για να μην υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις. για τα σημεία 26-28 μας είπε εκπρόσωπος του Εθνικού Συνεδρού κάποια πράγματα. Τα κρατημέλη του 26 θα μπορούσε να διαβάσει ο αναγνώστης. Δεν εφάρμοσαν ε, με τον τρόπο της απαιτήσει από ότι αυτή του σημείου 27 τα έκαναν λίγο καλύτερα και ακόμη πιο καλά τα έκαναν ε, οι χώρες του σημείου 28. Στα γενικά αποτελέσματα οι περιφέρειες, στις οποίες αναφέρεται στο σημείο 27, το ανεκτικό συνέδριο φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκή στον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν, ενώ άλλες ε, περιφέρειες, το 26, που ενώ διαβάζοντας εκεί δεν θα θεωρούσαμε ότι είχαν εφαρμόσει σωστά τα κριτήρια, τέλος πάντων για ε, τα πιο περιοριστικά, πούμε από τον πίνακα μετά ότι επαρκώς. Όχι υποδειγματικά, αλλά τέλος πάντων επαρκώς ε, υλοποίησαν ε, τα δέοντα. España solo por Cataluña o de, o de Alemania por Baden και να είναι αντίστοιχα αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή όχι μόνο όχι σε άλλες χώρες περιφέρειες και σε άλλες χώρες να είναι ολόκληρη η επικράτεια. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τις εκθέσεις, ασχολούμαι τώρα με τις του συνεδρίου, θα ασχοληθώ και στη συνέχεια. Ελπίζω, δεν ξέρω αν θα καταθέσετε τροπολογίες, ε, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη διοικητική διαδικασία. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Okay. Yeah. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και με το σημείο 5. Και συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο, ειδική έκθεση, διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγμένους οργανισμούς. Ινές. Έχουμε ακούσει ήδη μια παρουσίαση. Ήρθε η ώρα βεβαίως να ανταλλάξουμε απόψεις για το έγγραφο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. έχουμε να συζητήσουμε τα συμπεράσματα όχι μόνο της ε, διαδικασίας απαλλαγής των αποκεντρωμένων οργανισμών για πέρυσι και όλα αυτά τα οποία διδαχθήκαμε, αλλά είμαστε και στη φάση της ανάλυσης ενό σημαντικού στοιχείου, κριτηρίου δηλαδή της σύγκρουσης συμφερόντων, όχι μόνο στο πλαίσιο ορισμένων οργανισμών που αποτέλεσαν αντικείμενο και της έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου, αλλά και επειδή η Επιτροπή μας ε, πολύ σωστά αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο γενική προσέγγιση σε σχέση με ορισμένε πολύ σημαντικέ πτυχέ που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία και τη διαφάνεια τη διαχείριση του προπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όχι μόνο των αποκεντρωμένων οργανισμών, αλλά γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια ακρόαση και οι συστάσεις που περιλαμβάνουν και στην έκθεσή μου ε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσε. Θα μπορούσαν βέβαια να υπάρχουν και πολύ περισσότερες στάσεις. Να σας πω ότι ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά που μας δίδαξε η όλη ακρόαση και σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία θα τα βρείτε στην έκθεση του κ. Γκερμπράντι για την απαλλαγή σε ό,τι αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Εκεί δηλαδή αναφέρονται συγκεκριμένα αυτές οι πτυχές και μάλιστα ορισμένες βελτιώσεις ε, που επιλέξω όπως τις είχαμε ακούσει στην ακρόαση. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να διατηρούμε την διαφάνεια και την, την αυτονομία και ανεξαρτησία των επικεντρωμένων οργανισμών. Να λαμβάνουμε όμως υπόψη ταυτόχρονα και τις ειδικέ ανάγκες και σε περίπτωση διαχείρισης σύγκρουση συμφερόντων. Να βλέπουμε τις Άλλο είναι ε, ο οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και άλλο ο οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή ο Οργανισμός ε, ασφάλεια στη Θάλασσα ή ή τα θέματα διαχείριση εργασία. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. ό,τι αφορά τώρα τη στάση του ΩΣΑ για τις συμφερόντων. Τα έχουμε υπόψη μας, αλλά αφορούν πιο πολύ τις δημόσιες υπηρεσίες. Άρα δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επιχειρήσεων δημοσιοειδιωτικές. Ή αφορά τα διοικητικά συμβούλια. Εκεί έχουμε τις κατευθύνσεις γραμμές του ωσά που δεν καλύπτουν ε, το παιδί αυτό και χρειαζόμαστε ειδικού κανόνες. Χαιρόμαστε που μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, την περσινή, η Κομισιόν δημοσίευσε πλέον έναν οδικό χάρτη για την ανάγκη να έχουμε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για όλες τις πτυχές της σύγκρουσης περόντων δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Είδαμε ότι κάθε όργανο ανάλογα με τα προβλήματα δημιουργεί τη δική του διαδικασία και γι' αυτό χαιρόμαστε και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει αυτό το ρυθμιστικό πλάσιο, πλαίσιο πριν τα τέλη του 2013. Είναι σημαντικό οι κανόνες να μην πολλαπλασιάζονται, να μην ε, είναι σαν ζούγκλα, έχουμε δαχθεί ότι όσο πιο απλός είναι ένας κανόνας και δεν θα πει βέβαια απλός ότι δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα του τομέα στον οποίο εφαρμόζεται, αλλά ακριβώ. Επειδή κάποιος το σκέφτεται πάρα πολύ και ε, καταγράφει όλες τις ανάγκες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επεκταθεί. Πρέπει να αναφέρεται στις βασικότερες απαιτήσει, να είναι δηλαδή απλός ο κανόνας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι και αποτελεσματικό ο έλεγχος. Εάν είναι πολλές οι διακλαδώσεις, αν είναι πολύπλοκοι κανόνες, είναι δύσκολο μετά να ε, γίνει σωστά ο έλεγχος. Ούτε θα μπορέσουμε να πετύχουμε την απαιτούμενη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι γίνεται και μετά τις αρμοδιότητες των ε, τεχνικών, των ε, εμπειρογνωμόνων ή τι γίνεται με τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Έχουμε εδώ μια πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία, την Μεσολαβητή, που θα διερευνήσει αυτό το σύστημα, αν θέλετε, των περιστρεφόμενων θυρών. Για να δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πού είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Φυσικά οποιαδήποτε σχέση δεν συνιστά ε, αυτομάτως σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στον ορισμό και στην ταυτοποίηση αυτών των περιπτώσεων. Για να μην ε, τα συμπεριλάβουμε όλα και τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα σωστά κριτήρια. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το κομμάτι και νομίζω επίσης ότι αποτελεί πρόοδο το ότι μετά την έκθεση του Ανοιχτού Συνεδρίου και με τη νέα συζήτηση που είχαμε για την απαλλαγή το έτος 2011, είδαμε ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συνειδητοποίησαν την ανάγκη να αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων και έχουν προβήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις. Είναι σημαντικό το αναφέρει στην έκθεση του κ. Γκέρ Μπράντι. Πολύ καλά κάνει το ελεγκτικό συνέδριο και ελέγχει παρά Ακολουθεί την κατάσταση με τους οργανισμούς και ιδίως αυτούς που επηρεάζουν περισσότερο ό,τι αφορά προειδοποιήσεις για την υγεία και τα λοιπά, γιατί αυτές περισσότερο, αλλά γενικότερα. Καλό επίσης θα ήταν να έχουμε μια συστηματοποίηση, ώστε να έχουμε μια έκθεση για τη σύγκρουση συμφερόντων με διεύθυνση του πεδίου εφαρμογής. Καλό θα ήταν να δούμε επίσης ποιες, ε, ποιοι οργανισμοί υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί θα μπορούσαμε πιο αστερά να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η πανεξέταση του Μητρώου Διαφάνειας ε, και καλό θα ήταν ε, να βελτιώνεται μονίμως αυτό το Μητρώο. Τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα. Για τη διαφάνεια, για την δημοσιοποίηση των στοιχείων των ε, εμπειρογνωμών, των μελών, των διοικητικών συμβουλίων, τα βιογραφικά, τα, οι σχέσεις που έχουν, ε, τα συμφέροντα που έχουν κτλ. κτλ γιατί θέλουμε να έχουμε έλεγχο και διαφάνεια και τα πρακτικά των συνεδριάσεων ΔΔΣ θα πρέπει να δημοσιεύονται επίση. Όλα αυτά στο πλαίσιο των απαιτήσεων διαφάνεια, πρέπει να διατηρηθεί. Ξακολουθώ να πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρο των κινδύνων από τη σύγκρουση συμφερόντων έχει να κάνει με το ότι η Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση έχει γίνει πιο ευάλωτη, πιο τρωτή. Έχουμε τον κανονισμό υπηρεσικής κατάστασης, μείωση της εξωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων της Κομισιόν που είναι σημαντικό ελαχιστοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και της εξωτερικής ανάθεσης, γιατί αλλιώς έχουμε εκθετική αύξηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και δυσκολεύει και ο έλεγχος. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα βλέπουμε πολύ ε, σοβαρά όταν ε, ελαφρά την καρδία αποφασίζουμε να προβούμε σε εξωτερική ανάθεση κάποιων εργασιών της Κομισιόν. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς όταν στελεχώνουμε την Ευρωπαϊκή Διοίκηση με προσωπικό. Να μην πέσουμε ε, στην παγίδα του λαϊκισμού. Ότι δηλαδή κάθε υπάλληλο είναι πέραν οποιασδήποτε υποψία. Για να μην έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι έχουν συμφέροντα, συγκρούσει συμφέροντα, γιατί έρχονται από τη βιομηχανία και θα, πάνε, θα γυρίσουν στην βιομηχανία. Λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτούς τους υπαλλήλους με άλλους που δεν έχουν συγκρότηση συμφέροντα. Σίγουρα δεν πρέπει και να τους καταδικάσουμε σε, σε εξωστρακισμό από τη στιγμή που κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί να εξασφαλίσουν τα προστοζή με κάποιο τρόπο. Πρέπει να διδαχθούμε από τις δυσκολίες. Και πρέπει να ξέρουν το στομότερο δυνατόν υπάρχουν δυσκολίες για την εφαρμογή των ε, απαιτήσεων. Και αυτό να μας το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά να μας το λένε και αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Αυτά και περιμένω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ja, wollte Ναι, βλέπω ότι υπάρχει μία ερώτηση. Ο κύριος Μούλτερ που είναι εισηγητής για το επόμενο σημείο με έχει ενημερώσει ότι στις 5 πρέπει να φύγει και έχει μια άλλη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. Πρέπει όντως να παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό και ήδη έχουμε επεξεργαστεί το θέμα αυτό πολλές φορές ε, τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω σε αυτό το έγγραφο εργασίας να επαληθεύσουμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει το φύλλο πορείας της Επιτροπής. Γιατί λοιπόν να μην τους ζητήσουμε στην ετήσια έκθεσή τους να προετοιμάσουν μία συγκριτική, ένα συγκριτικό πίνακα με όλα όσα έχουν γίνει, όσα δεν έχουν ακόμα γίνει, όσα γίνονται και αυτά τα οποία δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για την υλοποίησή τους. Θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε και κάποιες δεσμεύσεις και να ζητήσουμε από τους διάφορους οργανισμούς όταν προετοιμάζουν τα προγράμματά τους και αυτό αφορά όλους τους οργανισμούς, όχι μόνο αυτούς που αναφέρονται εδώ στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, όλοι οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες να παρουσιάζουν ένα έγγραφο που να εξηγούν πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διαλέγουμε να κάνουμε ένα είδος δειγματοληπτικού ελέγχου. Τρεις παραδείγματος χάρη είναι υπηρεσίες, τρεις οργανισμοί, οι οποίοι να ελέγχονται όσον αφορά την υλοποίηση των ε, προγραμμάτων τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, έκθεσή σας. Είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό. Είναι πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιους ενιαίους κοινούς κανόνες όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων με ένα θέμα που προκύπτει πολλές φορές και σε πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εδώ επεξεργαζόμαστε σωστά, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι εμπερογνώμονες και οι ειδικοί, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η εργασία γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για κάποιον ιδιωτικό φορέα ή κάποια μεγάλη επιχείρηση. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτά που προτείνει στα συμπεράσματά σου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε όντως κοινέ κατευθυντήριες γραμμές, κοινού άξονες για τη δράση μας, αλλά θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ακριβώς ε, σύγκρουση συμφερόντων. Συγκεκριμένες ε, υποθέσεις όλοι κάνουμε, αλλά στην πράξη τι ακριβώς εμπίπτει σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει κάπου και στο κανονισμό του προσωπικού να υπάρξει αναφορά σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων γιατί ξέρετε ότι προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να εξαλείψουμε τις οποιασδήποτε επιρροές από μέρους ε, κάποιων κλάδων, κάποιων οικονομικών συμφερόντων, κάποιων επιχειρήσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που προτείνεις, αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να φτάσουμε σε ενιαίους κανόνες. Και όταν λέμε ότι βεβαίως κάποια από αυτά που μέχρι τώρα ίσχυαν θα πρέπει να πάψουν να ισχύουν, ε, αυτό είναι λίγο γενικό. Ας ξανακοιτάξουμε τα συμπεράσματα, ας δούμε πώς μπορούμε να τα εξειδικεύσουμε, να στοχεύσουμε τους τομείς τους οποίους θέλουμε να επεξεργαστούμε, έτσι ώστε να ισχύουν κάποια μέρα κοινοί κανόνες για όλους τους φορείς και για όλες τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια έκθεση πολύ σημαντική που φτάνει την κατάλληλη στιγμή. Στη χώρα μου ε, στα θέματα αυτά διαφθοράς και ε, συγκρούσεων συμφερόντων ε, περνάμε μία περίοδο αναταράξεων. Λοιπόν, πρώτον πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε απαλλαγή υπηρεσία και αναοργανισμό. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό από δημοσιονομικής απόψεως του ναντίον θα είναι δραματικό σφάλμα εάν η Κομισιόν ε, ζητήσει συνολική απαλλαγή. Δεύτερον, έφτασε η στιγμή να νομοθετήσουμε. Η έκθεση την οποία χαιρετίζω το υπογραμμίζει άλλωστε. Συμφωνώ με την ποιότητα των παρατηρήσεων της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, της συγγετρίας μας που έκανε μια τεράστια, ένα τεράστιο έργο. Τρίτον, θα πρέπει στην περίμετρο ελέγχου και εξέτασης να βάλουμε όλες αυτές τις δομές οι οποίες περιστοιχίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το Κοινοβούλιο βέβαια δεν συμφωνεί με τον υπερβολικά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει ε, όλες ε, τις ε, δομές οι οποίες περιστοιχίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις αναλύσουμε γιατί θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να καταλάβουν και οι διευθυντές και τα διοικητικά συμβούλια ότι πρέπει να υφίσταται τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Επίσης και ίσως η ομάδα μου δεν θα συμφωνήσει, αλλά εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, γιατί με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την ανεξαρτησία. Όταν ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιείται σωστά, αμείβεται καλά, ε, τότε υπάρχει ένα εχέγγυο ανεξαρτησίας. Ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια ε, ανεξαρτησία ε, και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς το, το κανονισμός το, της υπηρεσιακής κατάστασης Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Θα στραφώ προς την Επιτροπή. Έχετε κάτι να προσθέσετε σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομε παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα. Γιατί πραγματικά συμφωνεί με τις ανησυχίες μας και με τα σχόλιά μας στην Επιτροπή. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, είναι σαφής, πριν το τέλος του έτους θα υποβάλουμε κατευθυντήριες γραμμές και φυσικά θα πρέπει να τις επεξεργαστούμε από κοινού με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο έργο μας. Έχουμε ήδη υποβάλει ένα πρώτο σχέδιο στους διευθυντές των υπηρεσιών και φορέων. Έχουμε ξεκινήσει το διάλογο, περιμένουμε τις επίσημες αντιδράσεις τους. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ καλή η πρώτη αντίδραση. Καταρχήν λοιπόν όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να υπάρξει ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάγκη εμπειρογνωμοσύνης και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης, είναι σημαντικό να πει κανείς ότι αυτό που μας βοηθάει ιδιαίτερα το κύριο εργαλείο για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων είναι η διαφάνεια και βεβαίως η υλοποίηση των μέτρων που θα αποφασιστούν. Η κάθε υπηρεσία, ο κάθε οργανισμός θα πρέπει βεβαίως να αναλάβει τις δεσμεύσεις και όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, πολλά έχουν επιτευχθεί ήδη. Θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία των ε, φορέων αυτών και πιστεύουμε ότι πέραν αυτών των κατευθυντήριων γραμμών κάθε φορά που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή και υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Όμως πολύ σωστά είπε η κυρία Γιάλα ότι η αξιολόγηση κινδύνου σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων είναι αναπερίπτωση για την κάθε ε, υπηρεσία και τον κάθε οργανισμό διαφορετική και έχει δίκιο σε αυτό η συγκήτρια. Πολλά μέτρα θα πρέπει να υιοθετηθούν όπως ε, η δήλωση των ε, συμφερόντων, ενημέρωση, διαφάνεια σκοπός μας σε κάθε περίπτωση είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πριν το τέλος του 2013, να φτάσουμε σε μια κοινή προσέγγιση και βεβαίως, όπως λέμε και στο φιλοπορίες μας, θα συνεχίσουμε την ε, συζήτηση, το διάλογο και με την εισηγήτρια, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής ενδιαφέρεται για το θέμα και θα ήθελα να μας υποβάλει παρατηρήσεις αυτό. Ολοκληρώσαμε. Και το σημείο αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Γιατί πρόσθεσαν νέες ιδέες. που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο αυτού του εγγράφου εργασίας. έλεγχος εξολόγηση τη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να είναι ένας από τους πυλώνες και της δουλειάς Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σε σχέση με αυτό το οποίο σχολίασε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που θέλω και να τον ευχαριστήσω, Καλό θα ήταν βέβαια να δούμε και εμείς το σχέδιο που εκπονούν, και να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια. Απλά να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για την ευθύνη των οργανισμών και τον οδικό χάρτη. Εγώ είχα πει ότι με ανησυχεί κάτι. Πράγματι, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Και να είναι και ουδέτερο, όπως είπε και με στην Αλλά έχουμε δύο επίπεδα ευθύνης είναι αφενός υπεύθυνοι οι οργανισμοί άπαξ και έχουν θεσπιστεί τα κριτήρια, η φόρμουλα και οι διαδικασίες για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελικά η Κομισιόν είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους οργανισμούς. Δηλαδή, ναι, είναι ανεξάρτητη και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι οι οργανισμοί για να εφαρμόσουν και τις προτάσεις τους αλλά έχουν ε, και στο θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την Κομισιόν και, αυτές, και αυτοί οι οργανισμοί ευθύνη. Τώρα για τον οδικό χάρτη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό για, τις, ε, για τους επικεντρωμένους οργανισμούς, αλλά όταν πλέον θα έχει εγκριθεί το μέσο για τους οργανισμούς, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο διαχείρισης των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, και στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Διοίκησης, της Εκτελεστικής Επιτροπής υπάρχουν ειδικά προφίλ εξωτερικοί που εργάζονται σε πολύ λεπτά, για πολύ λεπτά θέματα και εκεί υπάρχει τόσο ο κίνδυνος να έχουμε σύγκρουση με κάποια εθνικά συμφέροντα. Και ξέρω γιατί μιλάω γιατί έχω υπάρξει εθνική εμπειρογνώμη. Όταν λοιπόν επιλύσουμε το πλέον επίγον που είναι ο δικός χάρτης για τη συγκρούσεις συμφέροντων των οργανισμών, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε λίγο ευρύτερα το θέμα και να καταρτήσουμε ένα γενικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή διοίκηση, τα διάφορα θεσμικά όργανα για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Έτσι πιστεύω θα εγγυηθούμε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κάτι που αυτή τη στιγμή, σε αυτούς τους ε, δύσκολους καιρούς, το χρειαζόμαστε. Όσο πιο αξιόπιστοι και διαφανεί είναι οι οργανισμοί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με εμπειρογνώμενε και ειδικού για, για τεχνικά ζητήματα. Το θέμα είναι να μπορούν οι πολίτε ε, να βλέπουν ποιο είναι ο καθένα και τι συμφέροντα έχει. Έτσι θα είναι και πιο καθαρές ε, από συμφέροντα ή αποφάσεις μας, πιο διαφανείς. Και θα μπορούμε να εξηγούμε στους πολίτες ε, και αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, είναι Σαγιάλα Σέντερ. Πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Μπορούμε να περάσουμε όμως στο επόμενο που είναι η αποστολή στο Καλίνγκραντ. Γιάν Μούλτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που ε, δεχτήκατε το αίτημά μου να ασχοληθούμε τώρα με το θέμα αυτό. Βεβαίως θέλουμε πολύ να επισκεφθούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον τμήμα της Ευρώπης. Δεν έχω πάει ποτέ μάλιστα εκεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ήδη έχετε ε, στη, στα στοιχεία που, στην τεκμηρίωση που έχετε. Το μόνο είναι θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν και από τις υπηρεσίες να μας δώσει όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα τις απαραίτητε πληροφορίες ε, γιατί είναι άγνωστο, αχαρτογράφητο περιβάλλον για μένα. Εάν τα στοιχεία για την παραχάραξη προϊόντων και για το λαθρεμπόριο σιγαρέτων, αν τα στοιχεία αυτά λέγω αληθεύουν, τότε πρέπει να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη πληροφόρηση από αυτόν. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, από το 1991 έχουμε δώσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε αυτήν την ε, περιοχή της Ευρώπης. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Θα, θα έπρεπε λοιπόν, ε, αν είναι δυνατόν, να μας δοθεί και ένας κατάλογος των προγραμμάτων ε, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν, δαπανήθηκαν τα κονδύλια αυτά. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να μας δώσει τον κατάλογο αυτό. Εγώ θα ήθελα, φτάνοντας στο Καλίνιγκραντ, να έχω όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες, έτσι ώστε να ξέρω και επιτόπου ποιες θα είναι οι πιο κατάλληλες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει κάποια νέα στοιχεία ή πληροφορίες. Τα ονόματα που έχω από μέρους της Επιτροπής είναι Κατάνια και Έγνουσπίλερ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε τις ετούμενες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μέχρι τώρα στην περιφέρεια του Καλίνιγκρατ έτσι ώστε να προετοιμαστείτε για αυτή την αποστολή. Επίσης ε, θα κάνουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία της, ε, του Καλίνιγκραντ έτσι ώστε να είναι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρόντες έτσι ώστε να συζητήσετε σαν αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα είμαι δυστυχώς ε, παρόν. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η αποστολή. Αλλά δυστυχώς έχω άλλες ε, οι κοινοβουλευτικέ υποχρεώσει. Θυμάμαι ότι παλιά είχαμε πάει ε, με την αντιπροσωπεία της ε, Ρωσίας, ε, τη οποία ήμουν πρόεδρο. Συζητήσαμε λοιπόν τότε για το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού. Είχαμε μάλιστα επισκεφθεί και την, το ίδιο σημείο διέλευση συνόρων που θα επισκεφτείτε τώρα. και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν και απαραίτητε συγκρίσει. Ευχαριστώ. Ποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο. κανεί, Θα ξαναδώσω τότε το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει. Κάποιος θέλει το λόγο. Α, από την Όλα θέλει κάποιος το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την πλευρά της Όλαφ Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή του Καλίνιγκραντ είναι πάρα πολύ σημαντική ε, λόγω ακριβώς ε, του μεγάλου αριθμού παράνομων σιγάρων. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές οι κατασχέσεις που έχουν γίνει, κυρίως της μάρκας Jin Lee, που παράγονται στην Ναπατκάια Φάμπρικα. Από στατιστική απόψεως να σα πω ότι το 2005 είχαμε ένα εκατομμύριο κατασχεμένα Jinling ε, τσιγάρα ενώ, ενώ το 2008 είχαμε φτάσει ε, στα 380 εκατομμύρια ε, τσιγάρα. Το 2011 το Gin Lin ε, Είχαμε μεγάλες κατασχέσεις αυτών των τσιγάρων δηλαδή στην ε, Λετωνία και στην Ουγγαρία, ε, στο δεύτερο μισό δε του ίδιου χρόνου και στη Γερμανία και στην Σλοβενία. Το πρόβλημα με το Jin Lin είναι ότι έχουν πλέον εδώ και 3-4 χρόνια κατακλείσει την γερμανική αγορά. Είναι καλής ποιότητα και χαμηλής τιμής. Επομένω, ε, η ε, διείσδυση στην αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική η πλευρά του ε, Καλίνιγκρατ ε, μετά από αίτημα αποσαφήνισης δικό μας ε, απεφάνθη ότι από τη στιγμή που τα τσιγάρα αυτά εξ αρχής φορούν ή προορίζονται μάλλον για εξαγωγή δεν, έχουν, δεν υπάρχει καμία παραβίαση αλλά το πρόβλημα ε, με, το με, τα, με τα, αυτά τα τσιγάρα gin είναι πολύ μεγάλο έστω και αν υπάρχει μία έτσι φθήνουσα πορεία. Η κυρία Γκρέσλε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι ρόλο παίζει το Καλίνιγκραντ για το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού. Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς. Υπάρχει, βλέπω κάποιους από την ε, Όλαφ και επιτόπου. Πολύ θα θέλαμε να το συναντήσουμε. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση κατευθείαν, κύριε Κατάνια. Ναι. Έχουμε μια συνεργασία και μια συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τις τελωνιακές αρχές, ε, βεβαίως και συνεργαζόμαστε στον τομέα αυτό και αναφερθήκαμε στις δύο επιχειρήσεις οι οποίες νόμιμα παράγουν προϊόντα jingling στην περιοχή του Καλίνιγκρατ. Πρόκειται για τσιγάρα τα οποία προορίζονται σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες καταρχήν και κατόπιν επανέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, την παράλληλη αγορά. Ναι, εγώ ζήτησα πληροφορίες την γραμματεία της Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης να έχουμε και την έκθεση που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια για το θέμα αυτό. Εγώ αναφερόμουν στην Επιτροπή, αλλά βεβαίως αν η Όλαφ έχει πληροφορίες, είστε ευπρόσδεκτη και με μεγάλη χαρά θα συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία και μπορείτε να μας υποβάλλετε οτιδήποτε έχετε θα είναι πολύ χρήσιμο για την αποστολή μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε και με το σημείο αυτό. Ολοκληρώνουμε και με το σημείο αυτό της μέσης διάταξης. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, την Όλαβ, Περιμένουμε τις πληροφορίες που μας υποσχεθήκατε για αυτήν την αποστολή. Νομίζω ότι αυτή η σύντομη ανταλλαγή απόψεων μας έδειξε ότι η αποστολή στο Καλίνιγκρατ έχει μεγάλη σημασία. Δικαιολογείται με το παραπάνω. Νομίζω ότι τελειώσαμε με τη δημόσια συνεδρίαση την σημερινή. Θα ξαναρχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 με το σημείο 9 τις ψηφοφορίες δηλαδή. Θα σε ευχαριστώ πολύ όλους. Οι συντονιστές μπορεί να παραμείνουν στην αίθουσα. Ξέρετε ποιοι αντικαθιστούν ε, ποιον. No. Okay. Υπάρχει αντικαταστάτης. Could you, could you, uh, Yeah. Ich, ich I propose that... Σας προτείνω λοιπόν να κάνουμε μια μικρή διακοπή, τρία με πέντε λεπτά και κατόπιν να συνεχίσουμε με τους συντονιστές. No. Mr. Skilakakis? I'm here. he is liberal, so... Yeah, I'm here. We'll arrive tomorrow.